σε ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Έχω και κάποιες άλλες ανακοινώσεις που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να σας πω ότι έγραψα στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για τα είδη διατροφή και οι λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας θα δημοσιευθούν στα πρωτόκολλα αυτής της ε, συνεδρίασης. Ο κύριος Χέρμουτ Σόλτ θα αντικαταστήσει